η διαδικασία του άρθρου 70α που είχα αναφέρει, θυμάστε ότι είναι μια νέα διαδικασία βάσει της οποίας οι συμφωνίες πρώτης ανάγνωσης μπορούν να εγκρίνονται από την Ολομέλεια. Για πρώτη φορά λοιπόν τίθεται σε εφαρμογή αυτή η διαδικασία και σας έχω φέρει τις προτάσεις της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για τα θέματα αυτά πρώτης ανάγνωσης. Μέσα στην προθεσμία που προβλεπόταν δεν υπήρξε καμία αίτηση για συζήτηση ή για ψηφοφορία. Επομένως, βάσει του άρθρου 70α, οι αποφάσεις αυτές θεωρούνται ότι έχουν εγκριθεί από την Ολομέλεια και θα ε, δημοσιευθούν στα πρακτικά της Ολομέλειας. Έρχομαι τώρα στη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης